Καλησπέρα σας. Επαναλαμβάνεται η σύνοδος. Έχετε τα πρακτικά τα χθεσινά. Υπάρχουν σχόλια. Περνάμε στην κοινή συζήτηση. για την κατάσταση στον αραβικό κόσμο, τη Βόρεια Αφρική, τη Συρία και την Ιεμένη μετά από δήλωση της Αντιπροέδρου και είπα της εκπροσώπου Βαρόνης Άστον που έχει αμέσως και το λόγο. Thank you very much, um, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Την περασμένη φορά που μίλησα εδώ στα τέλη Μαΐου είπα ότι δήλωση μπορούσα να κάνω και σωρό δηλώσει μπορούσα να κάνω, αλλά ότι η προτεραιότητα ήταν η δράση, η, τα έργα. Η ευρωπαϊκή σημαία βρίσκεται τώρα στην ε, νέο ονομαστήσα πλατεία της Ελευθερίας στη Βενγάζη ένα σύμβολο της αλληλεγγύης. Ε, το γραφείο μας ε, λειτουργεί και εμπειρογνώμονε καταφθάνουν κάθε εβδομάδα και δουλεύουν για να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις ε, ανάγκες ασφάλειας του λαού και να φτιάξουμε ικανότητε για την κοινωνία των πολιτών. Την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη συντονίζουμε τη εργασία με τον Ηνωμένα Έθνη για τη Λιβύη. Εμείς είχαμε επαφέ με ανθρώπους που αγωνίζονταν, αγωνίζονται για την δημοκρατία στη Λιβύη. Σας ευχαριστούν, με ευχαρίστησαν και ευχαριστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουν πως θα μείνουμε για αρκετό καιρό εκεί και είμαι βεβαία ότι και σήμερα θα θελήσετε να χαιρετήσουμε από κοινού το μέγα θάρρο του λιβικού λαού στη Βεγγάζη, στη Μιστράτα, στα Δυτικά Όρη ή αλλού. Εμείς έχουμε απειλήσει με κυρώσεις έχουμε δώσει 140 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια για να βοηθήσουμε αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο και εξακολουθούμε με επαφές. Θα έχουμε επαφή στην, στην Κωνσταντινούπολη αυτή την εβδομάδα και στην ομάδα του Κάιρο. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ κ. Αλχατή και τον ΟΗΕ, τον Αραβικό Σύνδεσμο αλλά και την ομάδα για τη Ισλαμική Συνεργασία. Προετοιμαζόμαστε για τι εβδομάδε και του μήνε μετά από την αποχώρηση του Καντάφη. Η δράση, βέβαια, θα πρέπει να βασίζεται σε στρατηγική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η πρώτη που σοβαρά απάντησε στην Αραβική Άνοιξη με την ε, ανακοίνωση τον Μάρτιο. Μετά δύο μήνες ε, ξεκινήσαμε μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική γυντνίαση και είμαι ευτυχής που έχω μαζί μου εδώ σήμερα τον, τον τον Στέφαν Φίλε που είναι ο στενός μου συνεργάτης σε αυτή την πολιτική. Γνωρίζετε ποιες είναι οι αρχές, αμοιβαία λογοδοσία, μεμονωμένες προσεγγίσεις στις μεμονωμένες χώρες ανάλογα με τις συνθήκες και τις προσδοκίες τους προσφορά μεγαλύτερη στήριξη για περισσότερε μεταρρυθμίσει. Για μεγαλύτερε Με τα λόγια του Στέφαν, more for more. Περισσότερα για περισσότερα. Επίση, έχουμε προβλέψει επιπλέον 1,2 δι ε, για τα επόμενα δύο χρόνια πάνω από τα πέντε ε, μάλλον ε, επιπλέον των 5 δις που ήδη έχουμε ε, δεσμεύσει, δηλαδή φτάνουμε στα 7,5-8 δις. Ξεκινήσαμε επίσης για να απεμπλακούν νέα επενδυτικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την ανοικοδόμηση και την αναδιάρθρωση και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όλα αυτά για την ενίσχυση της δημοκρατίας που θα ακολουθεί από την οικονομική ευημερία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η δημοκρατία δεν είναι σταθερή χωρίς ε, τρόφιμα, ασφάλεια και θέσεις απασχόλησης. Και τώρα αυτούς τους στόχους θέλουμε να επιτύχουμε. Πέρα από αυτή την πολιτική έχω αναλάβει δύο νέες πρωτοβουλίες από την τελευταία μας συνάντηση. Πρώτον για να ενδυναμώσουμε την πολιτική μας αποτελεσματικότητα, παρουσία και ορατότητα. Έχω ορίσει έναν μια νέα, ε, ένα νέο εκπρόσωπο για την Νότια Μεσόγειο, τον Μερναντίνο Λιόν, που έργο του θα είναι να ε, εμπλακεί σε διάλογο με τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους διεθνείς οργανισμούς και να συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερον, έχουμε φτιάξει μια task force ώστε να συγκεντρώσει τις δικές μας εργασίες και να ε, φέρει κοντά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την BERD, άλλους ε, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και διεθνείς εταίρους, ώστε οι δεσμεύσεις τους να μετατραπούν σε πραγματικότητα, να συγχρονιστούν και να συντονιστούν. Και αυτή η πραγματικότητα αφορά τη δημοκρατία και την οικονομία που θέλουμε να δούμε επί τόπου στην Τινησία και την Αίγυπτο. Βλέπουμε αποδείξεις των ε, αναταραχών τους τελευταίους μήνες. Πριν από λίγες μέρες που βρισκόμουν στην Αίγυπτο μίλησα με καταστηματάρχες, με ανθρώπους στον δρόμο, με ε, ξενοδόχους και όλοι μου λένε την ίδια ιστορία ότι τα εισοδήματα στον τουρισμό και στις άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν πέσει. Χρειάζονται στήριξη για να αναζωογονήσουν και να στηρίξουν την οικονομία τους. Γι' αυτό, για παράδειγμα, υποστήριξα μια μεγάλη πρωτοβουλία περί κοινωνικής ε, στέγασης στην Αίγυπτο ενώ στηρίζουμε έργα στην ευρύτερη περιοχή του Κάιρο καθώς και 20 εκατομμύρια πρόγραμμα για την κοινωνία των πολιτών της Αιγύπτου. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε την Αίγυπτο να μεταρρυθμίσει τον τομέα της ασφάλειας. Έχουμε προσφερθεί να στείλουμε αποστολή παρατήρησης και να βοηθήσουμε για την πορεία προς τη δημοκρατία. Έχουμε μιλήσει με τον Πρωθυπουργό Αλγαμάλ που ηγείται της προετοιμασίας των εκλογών, είναι εξέχον δικηνομικό και έχει αναλάβει το έργο να συντάξει το Σύνταγμα που θα είναι ο φύλακα του λαού. Επίση, την περασμένη Παρασκευή ήμουν στην Ισία όπου χρειάζεται στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και στήριξη επίσης για την προετοιμασία των εκλογών του Οκτωβρίου. Μας ζητήθηκε να στείλουμε αποστολή παρατήρησης των εκλογών και αυτό θα κάνουμε. Μεταρρυθμίσεις στην ασφάλεια επίσης ε, έχουν μπει σε κίνηση. Η κυβέρνηση της Τινησίας επίσης προωθεί τη δική της ατζέντα για τις μεταρρυθμίσεις και χειροκροτούμε τη συμφωνία που έγινε για την ημερομηνία των εκλογών και την αρχή ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών για τους καταλόγους υποψηφίων. Ανησυχώ για ολόκληρη την περιοχή ότι η φωνή των γυναικών θα πρέπει να συνεχίσει να ακούγεται και να είναι βέβαιη η συμμετοχή τους. Υπάρχει ένας φόβος που έχω ακούσει ότι αφού έλαβαν μέρος στην ε, Επανάσταση ε, η συμμετοχή τους στο μέλλον δεν είναι εγγυημένη. Θα πρέπει να το στηρίξουμε ε, με πόρους αλλά και από πολιτικής άποψης καταστώντας σαφές ότι περιμένουμε να τις δούμε μέσα στις εξελίξεις, στις μελλοντικές εξελίξεις. Στην Ισία θα πρέπει οι γυναίκες να συγκεντρωθούν το μικρόφωνο της ομιλήτριας διακόπηκε. Φυσικά μένουν πολλά ακόμη να γίνουν και παρεμπιπτόντως έδωσα σήμερα το πρωί μια δήλωση για την ανησυχία μου για τις πρόσφατες συλλήψεις γυναικών δημοσιογράφων. Ίσως όμως η μεγαλύτερη μας ανησυχία αναφορά το λαό της Συρίας που δεν που τους αρνούνται να ε, διεκδικήσουν τη δημοκρατία. Αυτό που ξεκίνησε ως τοπικές ε, διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς ε, στις τοπικές κοινωνίες έχει, γίνει, έχει μετατραπεί σε εθνική εξέγερση και έχει συναντήσει τη βία. 11 άνθρωποι πέθαναν μόλις 8. Πάνω από 500 πολίτες είναι νεκροί, 10.000 άνθρωποι κρατούνται αυτή τη στιγμή. Εμείς ε, καταδικάζουμε ανεπιφύλακτα αυτές τις βίες πράξεις. Από την τελευταία μας συνάντηση έχω αυξήσει τις κυρώσεις μας δις. Ε, συνεχίζω να μιλώ με τους διεθνείς μας εταίρους. Έχω αναζητήσει να ληφθεί δράση από το Συμβούλιο Ασφαλείας με στόχο να στείλουμε ένα μενιό μήνυμα, να σταματήσει η βία, να ξεκινήσει διάλογος και να γίνουν προετοιμασίες για την αλλαγή. Οι υποσχέσεις ε, του Προέδρου είναι αδύναμες, παραμένουν αδύναμες. Ε, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα θα συναντηθούμε για να προετοιμάσουμε το πλαίσιο του διαλόγου. Αλλά οποιοδήποτε διάλογος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Συμμετοχή δηλαδή της αντιπολίτευσης και όλοι όσοι συμμετέχουν να συμμετέχουν χωρίς φόβο. Η δική μας αντιπροσωπεία παραμένει επιτόπου στη Δαμασκό. Καθημερινά έρχεται σε επαφή με άτομα, ομάδες, δουλεύει με τους εκπροσώπους μας και στέλνει τα μηνύματά μας. Η αντιπροσωπεία μας στην Άγκυρα έχει επισκεφθεί πρόσφυγες που έφτασαν από τα σύνορα της Τουρκίας κατά χιλιάδες. Και εγώ ήμουν σε στενή επαφή με τον Πρωθυπουργό Νταβούτογλου της Τουρκίας για να προσφέρουμε ε, ό,τι χρειάζονται και αυτή η αστάθεια στην ε, Συρία φυσικά έχει απήχηση στον Λίβανο που βλέπουμε ειδικό, το ειδικό δικαστήριο ε, να συνεχίζει την εργασία του. Και εδώ ερχόμαστε στην αναζήτηση της ειρήνης ε, μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ. Οι αλλαγές στην γύρω περιοχή και η ομιλία του Πρόεδρου Ομπάμα, η κίνηση προς την Παλαιστινιακή συμφιλίωση, η προσεχής Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δίνουν νέα έμφαση στη δυνατότητα συνομιλιών και εξέβρισης λύσεις. Εγώ ακούραστα δουλεύω για αυτή τη δυνατότητα στενά συνεργάζομαι με τον πρόεδρο Αμπάς, με τον πρωθυπουργό Δανιάχου ε, και άλλους στην περιοχή σε συνεργασία με τις αραβικές χώρες ώστε να αναζητήσουμε έναν φιλόδοξο τρόπο να προχωρήσουμε όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίζει τον ηγετικό ρόλο όπως ακριβώς το επιθυμεί το Κοινοβούλιο. Ο ΙΕ, η ΙΠΑ και η Ρωσία απάντησαν στην, επιστολή μου για συνάντηση του κουαρτέτου και θα γίνει αυτό στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα. Έτσι θα συνεχιστεί η διαδικασία που ξεκίνησε στο Μόναχο με τις συναντήσεις, τη συνάντηση του κουαρτέτου. Έκτοτε οι επεσταλμένοι εργάζονται εντατικά και για πρώτη φορά με διαπραγματευτέ και από τι δύο πλευρέ. Δεν υποτιμώ την πρόκληση, αλλά στόχο μου είναι απόλυτα σαφή. Να βρούμε την επόμενη εβδομάδα έναν τρόπο ώστε να υιοθετήσουμε μια δήλωση που θα βοηθήσει του Ισραηλινού και του Παλαιστινίου να γεφυρώσουν τα κενά και να μπορέσουν να επιστρέψουν στη τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Πολλοί πρόεδροι προσβλέπουν στο Σεπτέμβριο και, προπτική, και στην προοπτική μιας, ε, ενός ψηφίσματος. Δεν ξέρουμε ακόμα τι μπορεί να λέει ένα τέτοιο ψήφισμα του ΟΗΕ και ποιες θα είναι αντιδράσεις σε αυτό. Αλλά είναι σαφές ότι η ενέργειά μας θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να κινηθούν οι συνομιλίες και γι' αυτό είναι ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε ε, μια πολύ ε, συμπαγή θέση από την οποία να κινηθούμε επί τη βάση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Επίσης καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τις ανησυχίες για το λαό της Γάζα. Έχω επισκεφθεί δύο φορές την περιοχή, έχω δει ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, η διεισόμαση και τονίζω με συνέπεια την ανάγκη να ανοίξουν τα σύνορα, οι σταθμοί, οι συνορικοί σταθμοί ώστε να παίρνουν τα αναγκαία οι κάτοικοι της περιοχής. Έχω μιλήσει και τα τελευταί, τις τελευταίες μέρες με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και γίνονται και επιτόπου επαφές, αλλά δεν υποτιμώ ότι πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν. Και ευχαριστώ την Ελλάδα ε, για την προσφορά της να στείλει διαθροπιστική βοήθεια στην Γάζα σε συνεργασία με τον ΟΗΕ. Να στραφώ τώρα σε δύο βασίλεια, στο Μαρόκο και στην Ιορδανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και ενθαρρύνει την δέσμευσή του για μεταρρυθμίσει. Στι 12 Ιουνίου, ο, King, ο βασιλιά Αμπταλά τη Ιορδανία διατύπωσε φιλόδοξε προτάσει σε σχέση με τα πολιτικά κόμματα και την εκλογική διαδικασία και είμαι σε τακτική επαφή με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τζουντέ, και στην τελευταία μου ε, επίσκεψη στην Ορδανία πριν δύο εβδομάδε. Είχα επαφέ εκεί και τέλο το τελευταίο Σαββατοκύριακο είχαμε καλά νέα από το Μαρόκο για τη μεταρρύθμιση του συντάγματο. Η μεταρρύθμιση αποτελεί ανταπόκριση στι θεμητέ ε, προσδοκίε του μαροκινού λαού. Ελπίζω πω οι μαροκινοί πολίτε θα παραμείνουν στο επίκεντρο τη διαδικασία εφαρμογή και ότι ο διάλογο τώρα θα διευρυνθεί και θα ενισχυθεί. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την πλήρη μας στήριξη στο Μαρόκο σε αυτή την προσπάθεια. Στην Αλγερία το... η κατάσταση επίγουσα ανάγκης έχει αρθεί και τώρα οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν στην πράξη. Όταν συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό της Αλγερίας το τόνισα αυτό. Και στον Παχρέιν Συνεχίζουμε να εκφράζουμε την ανησυχία μας για την συνέχιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα θυμάστε τις συζητήσεις με τον βασιλιά του Μπαχρέιν στον Περσικό κόλπο πριν λίγες εβδομάδες, αλλά ε, προσπαθήσαμε να ε, μιλήσουμε για την τροπιαστική συμπεριφορά απέναντι στους γιατρούς που προσπάθησαν να ε, βοηθήσουν όσους το χρειάζονταν καθώς και τα φρικτά που συμβαίνουν με την θανατική ε, ποινή εκεί. Ε, χρειάζεται να παραμείνουμε εκεί ισχυρή, ούτως ώστε να, συνε... να, επιτέλους να ξεκινήσει ο εθνικός διάλογος και τέλος να στραφώ στην Ιεμένη. Ακροτηριασμένη από το πολιτικό τέλμα και από τις επιδεινούμενες οικονομικές και ανθρωπιστικές συνθήκες, ο μόνος τρόπος που μπορούμε να προχωρήσουμε, όπως έχω συζητήσει με τον Πρόεδρο πριν να τραυματιστεί, και όπως ε, λένε τα μηνύματα που ξεκολουθούν να στέλνουν οι δικές μας αντιπροσωπείες είναι μια πραγματικά καθολική πολιτική μετάβαση σύμφωνα με τα όσα πρότεινε το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου στην πρωτοβουλία του. Εμείς συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας, το ΙΠΑ και το Συμβούλιο για να απεμπλακεί η κατάσταση και να βρεθεί λύση. Όσον αφορά ε, τον Πρόεδρο πρέπει να μεταφέρει την εξουσία του και να ακολουθήσει τη δέσμευσή του για μετάβαση. Εμείς έχουμε καταστήσει σαφέ ότι είμαστε έτοιμοι μαζί με τους διεθνείς μας εταίρους να δώσουμε περαιτέρω ανθρωπιστική πολιτική και πρακτική στήριξη. Αλλά δεν χρειάζεται να σας πω πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ιεμένη και πόσο Ανήσυχοι εξακολουθούμε να είμαστε λόγω των γεγονότων εκεί. Είμαστε επίσης έτοιμοι να βοηθήσουμε να προετοιμαστούν εκλογές και να, δι... να... να εγκαθιδρυθεί ένα λειτουργόν κοινοβούλιο. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για να λειτουργήσει η εμένη πρέπει να γίνει τώρα η μετάβαση. Πρόεδρε, να κλείσω ευχαριστώντας το κοινοβούλιο σα για την σταθερή του υποστήριξη για τις προσπάθειες διασφάλισης και προώθησης των θεμελιωδών δημοκρατικών αξιών, δικαιωμάτων και ελευθεριών. Το κοινοβούλιο αυτό είναι μοναδικό στα όσα μπορεί να προσφέρει σε όσα αναζητούν τη δημοκρατία. Εσείς είστε οι εκπρόσωποι της δημοκρατίας, αποδεικνύετε την, την, δύναμη των πολιτών, την ποιότητα της συζήτησης και της ελευθερίας έκφρασης. Πολλοί από εσάς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι προκλήσεις της οικοδόμησης δημοκρατίας, του αγώνα για ε, τα ιδεώδη. Έχετε πολλά να προσφέρετε στους, στους λαούς που έχω συναντήσει σε όλη αυτή την περιοχή, να, να πιέσετε για να αυξηθεί ο διάλογος και για τις ευκαιρίες να συναντηθείτε μαζί τους ώστε να βρεθούν πρακτικοί τρόποι ώστε να ριζώσει η δημοκρατία όπως ρίζωσε στις χώρες μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τους πείτε πώς ξεπεράσατε τις δυσκολίες. Ξέρετε πως θα είστε στην υποστήριξή σας για όσους ε, αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους προς τη δημοκρατία και προς το δικό τους μέλλον. Όπως μου είπε κάποιος ε, από τους πολλούς νέους που συνάντησα στη Βενγκάζη, ένας νεαρός ο οποίος ήταν στη φυλακή από τον Καντάφη ως πολιτικός κρατούμενος για 8 χρόνια, είπε «Θέλουμε αυτό που έχετε εσείς, δημοκρατία στην, σαν καθημερινότητα». Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτος μιλητής ο κύριος Σαλαφράγκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν τον Ορτέγα, έναν πολύ γνωστό διανοητή, τον ρώτησαν τι απόσταση πρέπει να πάρει κανεί από τα γεγονότα για να γράψει την ιστορία, είπε μία απόσταση όπου δεν μπορεί να ε, βλέπει κανεί ε, το περίγραμμα τη μύτη τη Κλεοπάτρα. Ε, Κυρία Άστον, αυτό σα το αναφέρω όχι γιατί η Αίγυπτο ε, έχει επηρεαστεί από την Αραβική Άνοιξη, αλλά γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο ιστορικό σταυροδρόμι. Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη ε, και πίστη ε, στο όραμά μα, κρίση χρέου, αμφισβήτηση των σημαντικών επιτευγμάτων τα οποία έχουν αναγνωρίσει οι πολίτε μα, όπω παραδείγματο χάρη είναι ο χώρο Σέγγεν, καθώ και αμφιβολίε για τι δυνατότητε του ΝΑΤΟ. Τα τελευταία όμω δυόμιση χρόνια έχουμε διαπιστώσει και αυτέ ε, βελτιώσει και αλλαγέ. Και εσεί που αναλάβατε τα καθήκοντα τη ΕΠΑΤΣ και αντιπροέδρου τη ε, Κομισιόν, ε, είχαμε επίση την ίδρυση τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, καθώ και την συνεργασία σε σχέση με την αναλωμένη πολιτική γειτονία. Και είπατε πολύ σωστά ότι οι γείτονέ μα πάντοτε θα βρίσκονται εκεί. Το θέμα είναι εμεί τι κάνουμε. Εμεί θα είμαστε στο ύψο των περιστάσεων θα είμαστε στο ύψο των προσδοκιών των πολιτών μας, οι οποίοι βλέπουν την εξωτερική πολιτική ως ένα ε, θερμόμετρο ε, που σφιγμομετρά την ευρωπαϊκή, τις ευρωπαϊκές ικανότητες. Θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις διαδικασίες μετάβασης στις χώρες που είναι αντικείμενο του ψηφίσματος που θα ψηφίσουμε αύριο. Εμείς σίγουρα, κυρία Άστον, είμαστε υπέρ όλων αυτών και θέλουμε και επιθυμούμε εσείς ε, να είστε επιτυχείς ε, στο έργο σας. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει μέγιστη δυνατή προβολή. Όχι, ε, δεν μιλάω για, το, για την προβολή και σε σχέση με αυτό που σας είπα πριν για τον Ορτέγα, αλλά πρέπει ε, να δείξουν, να, να βασιστούμε στον, ε, όχι στον ελάχιστο κοινοπαρονομαστή, αλλά στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμητή. Ευχαριστώ. Κυρία Ντεκάιζερ τώρα έχει το λόγο. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, έχετε εργαστεί πολύ και σίγουρα σας στηρίζουμε. Σας στηρίζουμε απόλυτα. Πάντως, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα αφορά χώρες που είναι λίγο λησμονημένες, δηλαδή Συρία, Μπαχρέιν, Εμένη. Και δίνοντας ε, εκεί έμφαση, ουσιαστικά ε, δύο στόχους έχουμε. Ο πρώτος στόχος είναι να πάψει η σιωπή και να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην περιοχή. Και οι χώρε που ανέφερα πραγματικά βιώνουν ε, ε, ματηρή καταστολή. Δεύτερο στόχο, ναι μεν παραμένουμε αποφασιστικοί, καταδικάζουμε του αποτροπιασμού που λαμβάνουν χώρα εκεί, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να αφήσουμε ένα πολιτικό χώρο για τι ενδεχόμενε διαπραγματεύσει. Και το ψήφισμά μα πρέπει να σα πω ότι το στηρίζουν ε, ευρέω οι διάφορε πολιτικέ ομάδε. Θα ήθελα να κάνω δύο-τρει παρατηρήσει μόνο. Η πρώτη είναι ίσως ανόητη, είναι γλωσσικού ε, περίχουμε. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη αραβικός κόσμος, αυτή η φράση. Δηλαδή τι υπάρχει ένας αραβικός κόσμος μόνο ε, όπως δείχνει το ψήφισμα, το είπατε και εσείς, υπάρχουν πολλές χώρες ε, με διαφορετικές ταυτότητες και χαρακτηριστικά. Υπάρχουν περιφέρειες, το Μαγκρέπ, το Μασρέκ και η ιδέα αυτή ενός αραβικού κόσμου νομίζω ότι κάτι πρέπει να ξεχάσουμε. Δεύτερη παρατήρηση, Συρία. Η καταστολή που σοβεί σε αυτή τη χώρα σήμερα είναι ε, ματηρή, είναι βίαιη, είναι ανελαίτη. Ε, ούτε τα παιδιά δεν γλιτώνουν από αυτήν και το ψήφισμα ε, καταδικάζει και καταγγέλει εγκλήματα τα οποία δεν μπορούν να παραμείνουν ατιμόρυτα και εκφράζει την ανησυχία για τα μεταναστευτικά ρεύματα, μάλλον τα ρεύματα προσφύγων. Πάρα πολλοί πρόσφυγες περνούν από την τουρκοσυριακή μεθόριο και ζητεί από την εθνική κοινότητα και από τον ΟΗΕ να παρέμβει. Καθώς επίσης ε, λέει και κάποια ε, πράγματα για σταθερότητα εντό και εκτό τη χώρα, αλλά δεν πάει πιο πέρα. Γιατί, παραδείγματο χάρη, γιατί δεν λέμε ότι θέλουμε ο Μπασάρ Ελασάντ να αποχωρήσει από την εξουσία από τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει το καθεστώ καταστολή, το οποίο από τον πατέρα. Δυστυχώ ο πρόεδρο αυτό έχει ε, υπερβεί τη διαχωριστική γραμμή και δεν υπάρχει επιστροφή. Θα πρέπει να γίνουν πολιτικέ διαπραγματεύσει ε, με τα χρώματα, αν θέλετε, τη Ευρώπη. Τώρα, η Συρία ξέρουμε ότι έχει, ε, έχει πνιγεί στη βία. Διάφορε μειονότητε θρησκευτικέ, κυρίω οι χριστιανοί, απειλούνται από εξτρεμιστέ, από ακραία στοιχεία δεν θα πρέπει να διστάσετε. Πρέπει να μεταβείτε στην Δαμασκό. Σα ζητώ, κυρία, ε, ε, είπατε εκπρόσωπο, αντίθετα από ό,τι υποπρολαλήσα σα συνάδελφο, εσεί να κρατήσετε μικρότερε αποστάσει. Πρέπει να υπάρχει ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία υψηλού επίπεδου. σω έχουμε ακόμα μια ευκαιρία. Σα παρακαλώ να προσπαθήσετε να την εκμεταλλευτείτε. Και τρίτη παρατήρηση γενικού περιεχομένου, επειδή περνάει, ε, τελειώνει και ο χρόνο μου, θέλω να πω ότι εμεί στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Έχουμε πολύ καλέ σχέσεις με αυτή την υπηρεσία, αλλά υπάρχει μια άλλη επικάλυψη ε, δομών, task force ε, και διαφόρων άλλων ε, φορέων. Πρέπει να παρασχεθεί η βοήθεια και η αρρωγή στις χώρες και θα πρέπει τα προβλήματα να τα ξεπεράσουμε. Και σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει και η ΕΕΔ και οι άλλες υπηρεσίες αυτές τις πολύ σημαντικές προκλήσεις. Ευχαριστώ. Κύριος δεν ξέρω αν είδατε τις τελευταίες ώρες και τις τελευταίες ε, μέρες ε, κάποια φιλμάκια στο YouTube. Εικόνες ε, που σοκάρουν. Ένας άνθρωπος στη Συρία που κινηματογραφούσε τις σκηνές, στους δρόμους και στα σπίτια και κάποια στιγμή όταν βλέπει ένα ελεύθερο σκοπευτή της προεδρικής στρατιωτικής φρουράς το σκοτώνουν, το σκοτώνει αυτός ο ίδιος άνθρωπος ε, που είναι ο ελεύθερος ε, σκοπευτής ε, που κινηματογραφείται. Αυτό που βλέπετε δηλαδή σε αυτό το φιλμάκι του YouTube είναι ο θάνατος του ίδιου του ανθρώπου που κινηματογραφεί. Και υπάρχουν πολλές τέτοιε περιπτώσεις. Ο άνθρωπος αυτός σκοτώθηκε γιατί προσπαθούσε να δείξει κάτι έπαιρνε εικόνες για να τις μεταφέρει στο διαδίκτυο και να μπορούν όλοι εκτός Συρίας να δουν τι συμβαίνει στη Συρία. Ούτως ώστε όλοι έξω από τη Συρία να μπορούν να δουν ότι συνεχίζουμε μετά από πάνω από 500 νεκρούς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε αυτή τη σφαγή και εμείς δεν κάνουμε τίποτα ή σχεδόν τίποτα για να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση. Ξέρω ότι η Συρία δεν είναι Λιβύη. Και δεν είναι στην πρώτη γραμμή της άμυνας. Αυτό το οποίο γίνεται στη Συρία είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο γίνεται στη Λιβύη. Και ίσως ακριβώς γι' αυτό η Συρία να είναι πιο δύσκολη περίπτωση στην αντιμετώπιση της. Όμω αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω από αυτό το οποίο τώρα κάνουμε. Και τι κάνουμε, περιμένουμε ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Βδομάδες τώρα περιμένουμε. Περιμένουμε και ελπίζουμε κάποια λύση με τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Κίνα για το θέμα αυτό, αλλά λύση δεν έρχεται. Επομένως το ερώτημα είναι όταν βλέπουμε live, όταν βλέπουμε ζωντανά τις σκηνέ επιτόπου, τις δραματικές αυτές σκηνέ. και από την άλλη μεριά βλέπουμε Βραζιλία, Ρωσία, Κίνα που τα μπλοκάρουν όλοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας ε, θα πρέπει ε, να σκεφτούμε κάποιο διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, να κάνουμε περισσότερα εμείς, αντί να περιμένουμε ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που δεν πρόκειται να έρθει νομίζω εγώ, κατά τις επόμενες μέρες ή και εβδομάδες. Έχω μια πρόταση γιατί νομίζω δύο πράγματα μπορούν να γίνουν. Αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε, επιπροσθέτω σε αυτόν που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, είναι πρώτον να επεκτείνετε τον κατάλογο των ατόμων ε, που αφορούν ε, οι κυρώσει. Μέχρι τώρα έχετε ένα κατάλογο 30 ετών σε συμφωνία με τι ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα Νομίζω ότι πρέπει να επεκταθεί ο κατάλογος στις 200 οικογένειες που βρίσκονται στην εξουσία στη Συρία αυτή τη στιγμή και που συνεχίζουν να υποστηρίζουν τον Ασάντ και κερδίζουν χρήματα χάρη στο καθεστώς. Νομίζω ότι πρέπει να επεκταθεί ο κατάλογος γιατί ο Ασάντ βρίσκεται ακόμη στην εξουσία χάρη σε αυτές τις 200 οικογένειες και η σφαγή συνεχίζεται χάρη σε αυτές τις 200 οικογένειες. Και χάρη σε αυτές τις 200 οικογένειες υπάρχουν τέτοιοι ελεύθεροι σκοπευτές σαν αυτόν που είδατε στο διαδίκτυο, στο φιλμάκι αυτό του YouTube, που σκοτώνουν ανθρώπους ανθρώπους στους δρόμους. Δεν μπορούμε να κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια και να περιμένουμε επί εβδομάδες ένα ψήφισμα των εθνών που δεν φτάνει. Θα πρέπει να ε, επεκτείνουμε την απαγόρευση ε, ταξιδίου και ε, και στις 200 αυτές οι οικογένειες που ανέφερα που υποστηρίζουν τον Ασάντ. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει κυρία Άστον. Γιατί πρέπει τελικά να δούμε την πραγματικότητα δεν υπάρχει πρώτη γραμμή άμυνα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο όπως στη Λιβύη. Αλλά τουλάχιστον να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τη δυνατότητα δημιουργίας μέσα στη Συρία μιας ασφαλούς ζώνης. Μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μέσα στο έδαφος της Συρίας και αυτό δεν είναι ευσεβισπόθη, διότι στην Άγκυρα αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο κατεργάζονται. Αυτό σκέφτονται. Το 1991 στο Ιράκ έγινε ήδη με την υποστήριξη των ΗΠΑ για να προστατευθούν οι πολίτες που ζούσαν στο βόρειο τμήμα του Ιράκ και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε να βλέπουμε να συμβαίνουν αυτά τα οποία μόλις σας περιέγραψα, όλο και περισσότερες ε, ε, σφαγές. Η πρότασή μου λοιπόν είναι να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση γιατί δεν πρόκειται να έχουμε ομοφωνία στα Ηνωμένα Έθνη και δεν θα έχουμε ψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Πρόεδρε, ο εκπρόσωπο μας, ε, έξι μήνε μετά την ε, ε, έναρξη της Αραβικής άνοιξη, συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Χρειάζεται να επενέσουμε την Αίγυπτο γιατί οδήγησαν στο δικαστήριο τον Μουμπάρα και την οικογένειά του. Η πολιτική μας ομάδα, το ECR, ελπίζει ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε ένα νέο πρόεδρο στην Αίγυπτο που θα μπορέσει να αποκαταστήσει το γόητρο της ε, ε, Αιγύπτου. Και πρέπει να πω εδώ ότι ο αραβικός κόσμος υπάρχει και μπορούμε να συνεχίσουμε τον αποκαλούμε αραβικό κόσμο. Ε, η Αίγυπτος συνέχισε τις συμφωνίες ειρήνης με το Ισραήλ και αυτό είναι σημαντικό βήμα για την ειρήνη. Ε, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Λέδη Άστον όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ανασυγκρότηση και ανάπτυξη ε, και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ε, Επενδύσεων. Και η Τινησία συνεχίζει να κάνει πρόοδους προς ένα πιο σταθερό μέλλον, παραμένει όμως αποσταθεροποιημένη από τις εξεγέρσεις στη γειτονική Λιβύη και είναι σημαντικό για την αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ που Βάλει το ψήφισμα 1973 των Ηνωμένων Εθνών να σταματήσει η κατοχή του Καντάφη στην ε, Λιβύη. Εμείς στη Δύση δεν μπορούμε να αφήσουμε μισοτελειωμένη τη δουλειά ε, στη Ρωσία γιατί ένας τραυματισμένο Καντάφη που θα του επιτραπεί να παραμείνει στην εξουσία θα είναι καταστροφή γιατί θα προσπαθεί να εκδικηθεί έναντι των δικών του των ανθρώπων. Επίση, θα έπρεπε να αναφέρουμε και την ε, Αλγερία που ε, ε, συνεχίζει να υπάρχει πέρασμα μισθοφόρων από την Τρίπολη και ο βασιλιάς Αμπτουλάχ είναι τμήμα του προβλήματος ε, και όχι της λύσης. Παρακαλούμε λίγο πιο αργά, λέει ο πρόεδρος. Θα σας δώσω λίγο περισσότερο χρόνο. Καταλαβαίνουν όλοι αγγλικά, λέει ο κύριος Τάνοκ. Δεν πειράζει που το προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Θα σας δώσω περισσότερο χρόνο, λέει ο πρόεδρος, αλλά αν μπορείτε λίγο πιο αργά γιατί δεν μπορούν να μεταφράσουν οι διερμηνείς. Έλεγα λοιπόν ότι είναι τμήμα του προβλήματο και όχι τη λύση ο βασιλιά Αμπτουλάχ και πρέπει να μείνει στην ε, ε, Σαουδική Αραβία και να ετοιμάσει ε, την κατάσταση για του διαδόχου. Ναι, και στο Μπαχρέιν η κατάσταση ανησυχητική γίνονται κάποιες παραχωρήσει έναντι της αντιπολιτευτικής πλειοψηφίας των Ασία. Και ε, δεν μπορούμε να ξεχνάμε την ε, κατάσταση στη Συρία. Ε, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται που ζητούν μια δημοκρατική Συρία χωρίς την αρνητική επίπτωση της επιρροής του Ιράν. Μα, μας ανησυχούν οι ανακοινώσεις ε, για ε, ομάδες ε, που ενώνονται με τους πολίτες που διαμαρτύρονται και ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχουν προπαγανδιστικέ κινήσεις. Επίση, χαιρετίζουμε τι συνταγματικέ μεταρρυθμίσει στο Μαρόκο για να μειωθούν οι εξουσίε του βασιλιά και η κατάσταση στην Δυτική Σαχάρα μπορεί να επιληθεί με ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία. Την περασμένη εβδομάδα χαιρετήσαμε το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του, του Σουδάν και δεν θα πρέπει πρέπει να αποσταθεροποιηθεί το πιο νέο έθνος της ε, Αφρικής στην νέα αυτή προσπάθεια. Ευχαριστούμε για όλη την καλή σας δουλειά και για την υποστήριξή σας για την υποστήριξη της Αραβικής ε, Άνοιξης και για τη σταθεροποίηση των γειτόνων μας προς νότων. Ευχαριστώ κυρία Φλότχ. Σας ευχαριστώ. Είμαι τεράστια ενέργεια που χρησιμοποιούν οι αραβικοί λαοί αυτή τη στιγμή για να ανατρέψουν τα καθεστώτα που του τους ε, καταπιέζουν και καταρρύπτει πολλά από τα όσα πιστεύαμε για τους, την αδράνεια και την απάθεια των ε, Αράβων. Επίσης έτσι εξαλείφονται οι διάφορες συμφωνίες που είχαν συναυθεί με τις ε, ξεπερασμένες αυτές εξουσίες, καταργούνται οι τυραννίες. Θα πρέπει να σταματήσουν όμως οι απόπειρες ε, καθοδήγηση των επαναστάσεων αυτών. Θα πρέπει να δουλέψουμε με τάρρους που θα λογοδοτούν πλέον απέναντι στους πληθυσμούς τους μια πραγματική ε, ε, επανάσταση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος πιστεύει σήμερα πως ο Μπασάρα Λασάν θα μπορέσει να ξεκινήσει μια πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε εκδημοκρατισμό. Εγώ πάντως σίγουρα δεν το πιστεύω αυτό και ούτε και πολλοί κόσμος το πιστεύει. Εν πάση περιπτώσει αυτή η έκκληση να εγκαταλείψει την εξουσία Μπασάρα Λασάντα δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και πλειοψηφία για να χαρακτηρίσει τις βιότητες, ε, τις φρικαλαιότητες αυτού του καθεστώτος ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γιατί περί αυτού πρόκειται και να απαιτήσει μέσω ενός ψηφίσματο του Συμβουλίου Ασφαλείας την ε, οδήγησή του στο Διεθνές ε, Ποινικό Δικαστήριο. Νομίζω πως ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το επιχείρημα για τις διστακτικές χώρες, τη Ρωσία και την ε, Κίνα, καθώς και τη Βραζιλία. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η προστασία η προσωρινή, να υπάρξει βοήθεια στην ε, θάλασσα. Αυτό να προτείνει στους πρόσφυγες ο ΙΕΒ και όχι να διοργανώνει ε, συνεδριάσεις κρίσης. Ε, αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ε, που θα εγγυάται τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις φάσεις για την ε, εκπόνηση των πολιτικών, για την αξιολόγηση των δικτών, τη συνεργασία με του μελλοντικού μα εταίρου, γιατί η πραγματική αλλαγή εκεί έγκυται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κοινωνικοί εταίροι που θα, θα λογοδοτούν ενώπιον των πληθυσμών του και εκείνοι ε, οι πληθυσμοί διψούν για εκδημοκρατισμό. Σωστά τα αναλύσατε, κυρία Άστον. Πριν από τις, την Επανάσταση, στην αρχή τη εντολή σα, είπατε ότι η αξιοπιστία τη εξωτερική μα πολιτική ε, παίζεται στην ε, γειτονία μα, την άμεση, και είχατε δίκιο. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για δημοκρατία στους λαούς μας, δεν θα, είμαστε, δεν θα πρέπει πια στην, να ενεργούμε με ερωτηματικά, αλλά να μιλάμε για το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τον 21ο αιώνα. Αυτό διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ματίας. Κυρία Άστον, εγώ ξεκινώ Λέγοντα πώ είναι προφανέ ότι οφείλουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τι δημοκρατικέ επαναστάσει που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη χώρα. Δεν έχω πολύ χρόνο και γι' αυτό θα ήθελα μόνο να σα πω δύο λόγια. Καταρχήν, ε, μπορούμε να πούμε ότι οι προποθέσει για να υπάρξει εκδημοκρατισμός και όχι φίλος πόλεμος θα πρέπει να καθοριστούν από τους ίδιους τους χώρους που διαμένουν στις χώρες. Η κατάσταση στη Συρία είναι πολύ σοβαρή ε, πολύ κρίσιμη και αν θέλουμε να αποφύγουμε τον εμφύλιο πόλεμο, τελευταία που ε, χρειάζονται οι χώρες αυτές είναι να ανακατεύεται η Ευρώπη στα εσωτερικά τους κυρίως υποβάλλοντας ε, στρατιωτικές, προτείνοντας μάλλον στρατιωτικές ή παραστατικές λύσεις. Και αυτό το λέω γιατί θέλουμε να αρνηθούμε τα όσα γίνονται στη Λιβύη. Το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι έχουν ξεπεράσει κάθε ψήφισμα, ακόμα και αυτά που ψήφισε το Συμβούλιο Ασφαλείας της, του, του Και αυτή η σιωπή απέναντι στη Λιβύη είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται και με αυτό εδώ το ψήφισμα και εγώ τουλάχιστον δεν θα το υποστηρίξω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέλντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 ο Μπεν Κουριόν, ιδρυτής του Ισραήλ, έλεγε, έλπιζε ότι θα μπορούσε να ε, υπάρξει ένα άνοιγμα με την αλληλή καθισότητα του Ισραήλ, ένα άνοιγμα προς ε, τους αραβικούς λαούς. Και υπήρχαν άλλοι, ε, όπως το καθεστώς Νάσερ και άλλοι, που ήταν ακόμη πιο ε, από ε, τους μονάρχες οι οποίοι εξέπεσαν της εξουσίας τους. Εγώ ε, θέλω να πω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε να υπάρξει ε, παραλληλισμός με τη δεκαετία του 50 σήμερα στην Αίγυπτο. Ξέρουμε ότι η μουσουλμανική αδελφότητα επηρεάζει, προσπαθεί να μπλοκάρει οποιαδήποτε ειρήνευση με το Ισραήλ. Πρέπει να υπάρχει πιο θετική στάση. Πρέπει να βελτιωθούν οι Ισραηλινο-αραβικές παλαιστινιακές σχέσεις. Ο Ελ Μπαραντέι, ο Άμπρε Μούσα που είναι ε, πιο συμφιλιωτικοί ε, δεν βλέπω να δημιουργούν ε, εμπιστοσύνη στο κράτος του Ισραήλ. Η... Το Ιράν επίσης απειλεί να καταστεί ένας πραγματικός εφιάλτης σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο για την περιοχή αυτή. Πώς μπορούμε και με την συνεργασία των ΗΠΑ ένα τέτοιο σενάριο να το αποφύγουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μάλτσερ. Κύριε Πρόεδρε, για πολλές αραβικές ε, χώρες ε, δεν υπάρχει γυρισμός σε σχέση με αυτά τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν. Ε, υπάρχει κάποια ελπίδα και για το λαό της ε, Ιεμένης ε, όταν βλέπουμε το λαό που αγωνίζεται. Δεν θα αλλάξουν και πολλά με μια αλλαγή προέδρου όπως προβλέπεται από το Συμβούλιο του Αραβικού Κόλπου. και τα προβλήματα συνεχίζονται όπως βλέπουμε και στις επιθέσεις που γίνονται στην Αίγυπτο κατά των ε, χριστιανών. Τα προβλήματα ε, ασφαλείας, τα ε, προβλήματα της οικονομικής κατάστασης είναι κάτι το οποίο οφείλεται στα παλαιά καθεστώτα. Και μετά το Μαρόκο και στις άλλες χώρες ε, ε, ξέρουμε ότι υπήρξαν ε, περιστατικά έντονης βίας. Αν μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση, πιστεύω ότι θα είναι και η Συρία ευεργετικό Ξέρουμε ότι υπάρχει από την κατάσταση αυτή στις αραβικέ χώρες ο κίνδυνος ροή νέων προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό ε, θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε ε, υπόψη για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε μελλοντικά προβλήματα. Ευχαριστώ και εδώ κλείνω ο κατάλογο των ομιλητών από τις πολιτικέ ομάδε. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ μια αντιπροσωπεία από την Βουλή της Βραζιλίας, η επενδυσία του Κάλλος Αλβέρτο Λαρέα, που βρίσκονται στο θεωρείο. Παρακολουθούν την συνάντηση Κοινοβουλίων Ευρωπαϊκής Ένωσης Βραζιλίας, που είναι